τα πλήρη δικαιώματα των ευρωβουλευτών και συμμετέχουν στη συνεδριά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε τα διαπιστευτήρια των, ε, της κυρίας Άλεξ Μαϊερ και του κυρίου Τίμο Βέλκεν και κύρωσε τις έντολες τους ε, από 15 Νοεμβρίου και 14 Νοεμβρίου 2016 αντιστοίχως. Υπάρχουν αντιρρήσεις.